Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir euh, nos travaux. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Είχαμε φτάσει μέχρι το σημείο 8. Θα εξετάσουμε δηλαδή τις ε, τροπολογίες της έκθεσης της Ελιζαμπέτ Σρέντερ, που είναι έκθεση πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας. 136 τροπολογίες έχουν κατατεθεί για την έκθεση αυτή. Βλέπετε το τεράστιο φάσμα συζήτησης υπάρχει. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για το μεγάλο σας ενδιαφέρον και τις και οι πολλές τροπολογίες γενικά αποτελούν βελτίωση, υπάρχουν κάποιες διαγραφές. Όλοι όσοι ήταν εισηγητέ ε, γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να μην προκαλεί πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά όλες οι υπόλοιπες ε, τροπολογίες αποτελούν βελτίωση του κειμένου ως προς το περιεχόμενο και προσπαθήσαμε στο γραφείο μου να τις συνδυάσουμε, δηλαδή να βρούμε ε, συμβιβαστικές τροπολογίες για τις μεμονωμένες παραγράφους ε, που να περιλαμβάνουν στοιχεία από τις μεμονωμένες αυτές τροπολογίες. Επιπλέον, πέντε επιτροπές ε, γνωμοδοτούν ε, έχουμε πάνω από 60 τροπολογίες από αυτές. Οι περισσότερες επιτροπές ε, ήδη ψήφισαν, ε, τις παρακολουθήσαμε και έχουμε κάνει κάποιους προσωρινούς καταλόγους σχετικά με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Μία επιτροπή λείπει ακόμα, η Ήτρε που είναι σημαντική επιτροπή και που έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες. Θα υπάρξει λοιπόν ε, και εκεί σημαντική συνεισφορά ως προς το περιεχόμενο. Και γι' αυτό είπα στους σκιώδεις εισηγητές ότι δεν μπορούμε ακόμα να υποβάλουμε συμβαστικές τροπολογίες, γιατί πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από την Ήτρε για να καταλήξουμε σε ε, κάποιον συμβιβασμό όσον αφορά την ενέργεια, τη βιομηχανία κλπ. Γι' αυτό περιμένω λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Υπολογίζουμε λοιπόν ε, είτε αυτή τη βδομάδα είτε το αργότερο τη Δευτέρα να έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες ε, τις οποίες θα στείλω στους σκιώδεις συζητητές ώστε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε το χρόνο να τις εξετάσουμε, διότι σίγουρα είναι πολλές. Παράλληλα, ε, με κάποιους ε, που έχουν υποβάλει τροπολογίες ε, και με τους οποίους υπάρχει προφορική συμφωνία. Έχω λάβει απαντήσεις από κάποιους από αυτούς. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα, εκκρεμούν ακόμα τα ζητήματα. Οι σκιώδεις εισηγητές και αυτοί που έχουν υποβάλει τροπολογίες ξέρουν ότι ανα πάσα στιγμή είμαι στη διάθεσή τους. Ε, μπορούμε λοιπόν να έχουμε διμερείς διαπραγματεύσεις. Ε, είμαι κατά των διαγραφών και είμαι κατά της τροποποίησης τίτλων, διότι πιστεύω ότι έχουμε ε, εντολή. Η έκθεση πρωτοβουλίας εγκρίθηκε με το συγκεκριμένο τίτλο και θα ήθελα να μείνω σε αυτό με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ε, σας απαριθμίσω όλες τις ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι η γραπτή διαδικασία είναι πιο κατάλληλη. Merci. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ουσάγια και μετά ο κύριος Λουτβίξον. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Liityn näihin Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για τις τροπολογίες που κατέθεσε που είναι πολύ επικοδομητικές και βελτιώνουν την έκθεση. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ σε κάποιες προτάσεις των τροπολογιών 1 ως 7. Εγώ υπέβαλα αυτές τις μνήες στις εν λόγω τροπολογίες, γιατί ήθελα να αποκαταστήσω κάποια ισορροπία. Στις ε, τροπολογίες 10 έως 13 εξετάσαμε το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας αλλά και τις επιδοτήσεις, τα θέματα της φορολογίας και, τα... και τις άμεσες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για τις προσλήψεις. Η χρήση αυτών των επιχορηγήσεων θα πρέπει να γίνει με βάση μελέτες, έρευνες. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε αρκετά διεξοδικές μελέτες για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση που κάνουμε αυτών των επιχορηγήσεων. Θέλουμε όλοι σίγουρα περισσότερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη ανάπτυξη, ευημερία και ελπίζω αυτή η νέα στέρη οικονομική βάση να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Βέβαια, δυστυχώς οι χώρες είναι υπερχρεωμένες, έχουν υπέρογκα δημόσια χρέη και είναι σε ευάλωτη θέση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δούμε τι επιχορηγήσεις θα χρησιμοποιήσουμε, τι φορολογικά μέσα και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Χρειαζόμαστε μια σφαιρική, ε, ολιστική οικονομική προσέγγιση. Είμαι υπέρ μιας σφαιρικής προσέγγισης από οικονομική άποψη. Επίσης, ε, στις ε, τροπολογίες 14, 15 και 16 μιλάμε αρκετά για τις ε, εργασιακές συνθήκες. Πιστεύω ότι με μια προφορική τροπολογία θα βρούμε μια καλή συμβαστική λύση. Εμείς στις σκανδιναβικές χώρες έχουμε γενικές συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους. Και δεν νομίζω ότι είναι χειρότερη ποιότητα αυτών των θέσεων εργασίας. Με τις συλλογικές συμβάσεις εξασφαλίζουμε τις ίδιες εργασιακές συνθήκες και στις νέες θέσεις απασχόλησης, αντίστοιχες με αυτές που ίσχυαν για τις παλιότερες. Θα ήθελα να μιλήσω για τις τροπολογίες τώρα 54 έως 63. Εκεί μιλούμε για τις ποσοστώσεις. Εγώ προέρχομαι από σκανδιναβική χώρα. Είμαι υπέρ της ισότητας των φύλων. Δεν νομίζω ότι οι ποσοστώσεις είναι το ιδανικό μέσο για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών στον χώρο εργασίας. Αντίθετα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ισότιμες προϋποθέσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες και στα θέματα επιμόρφωσης και κατάρτισης. Εγώ δεν είμαι υπέρ των ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, στις ηθήνουσες θέσεις κτλ. Τώρα, τροπολογίες 92 έως 104. Ε, Αναφέρεται η φορολογία Τόμπιν εδώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη νέα οικονομική κατάσταση και αν δημιουργήσουμε νέους φόρους, αν θεσπίσουμε νέες μορφέ φορολογίας, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί και να εκπονήσουμε μελέτες πριν θεσπίσουμε νέα φορολογικά μέτρα ή νέους φόρους, ακόμη και για τη φορολογία Τόμπιν. Θα πρέπει να κάνουμε διεξοδικότατη μελέτη για τις επιπτώσεις ε, ενός τέτοιου νέου φόρου πριν κάνουμε το βήμα της θέσπισης του. Τέλος. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία για την έκθεση, αλλά και σε συμφωνία για τις φιλοπεριβαλλοντικές θέσεις απασχόλησης. Βέβαια στις τροπολογίες χρησιμοποίησαμε διαφορετικούς όρους άλλοτε λέμε πράσινε θέσει εργασία και άλλοτε βιώσιμε θέσει εργασία. Θα πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία και να χρησιμοποιούμε έναν ενιαίο όρο. Προτιμώ να χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο και εγώ προτιμώ το βιώσιμε θέσει εργασία από το πράσινε. Γιατί αλλού αναφέρεται το ένα και αλλού το άλλο και αυτό δημιουργεί σύγχυση. Για μένα το green jobs είναι πιο πολιτικοποιημένη έννοια από το βιώσιμε θέσει απασχόληση. Ναι, μιλούμε για πράσινες θέσεις εργασίας, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πράσινες και αξιοπρεπείς. Ο κύριος Λούντβιξον και μετά ο κύριος Σταμασμάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή της έκθεση. Εξέτασα τις τροπολογίες ε, και είδα και βελτιώσεις και τροπολογίες με τις οποίες δεν συμφωνώ. Υπάρχουν επίσης ε, τροπολογίες τις οποίες δεν καταλαβαίνω, όπως για παράδειγμα τη διαγραφή στην αναφορά των μακροπρόθεσμων πλαισίων, κάτι που χρειάζεται η βιομηχανία για να μπορεί να προγραμματίσει χωρίς ε, πολλούς παράγοντες ε, ανασφάλειας. η βιομηχανία χρειάζεται μακροπρόθεσμα πλαίσια. Ξέρει κανείς λίγο πολύ τι θα συμβεί. Πρέπει να γνωρίζει κανείς περίπου τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια για να μπορεί να προγραμματίσει την παραγωγή του. Και ε, για αυτού τους νέους τύπους ε, θέσεων εργασίας θα πρέπει να χρειάζεται μακροπρόθεσμα πλαίσια. 136 τροπολογίες υπάρχουν ε. και υπάρχουν πολλές παρόμοιες προτάσεις. Κάποιες είναι πιο επικοδομητικές από άλλες φυσικά, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχουν καλοί λόγοι να συνεχιστεί η συζήτηση και προσλέπουμε στην συζήτηση των συμβιβαστικών τροπολογιών, την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουμε λάβει και τις νομοδοτήσεις των άλλων επιτροπών. Βρίσκω πολύ θετικό το να μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμούς επειδή είναι σημαντικό το θέμα αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε ευρεία στήριξη της πρότασης αυτής. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Λούτβιξον. Πολλά δε μάλλον που ήσασταν και λακωνικό. Ο κύριο Τόμα Μάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Ελίζα Περσρόντερ όχι μόνο για την έκθεσή τη, αλλά και για το ε, γεγονό ότι είπε ότι θέλει να έχει ενεργή συζήτηση όχι μόνο με τους σκιώδει εισηγητέ. Έχω υποβάλει και εγώ τροπολογίες. Πιστεύω ότι σε πολλούς τομείς θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Μία ερώτηση έχω όσον αφορά την ποσόστοση για τις γυναίκες. Ε, η Ζάρη το ανέφερε αυτό ήδη στην πρόταση αναφέρεται ποσόστοση γυναικών 40% ε, στις διοικήσεις επιχειρήσεων. Ε, στη Γερμανία ε, η νέα υπουργό είπε ότι θα πρέπει να έχουμε ποσόστοση. Άλλοι πολύ σωστά είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε ποσοστώσεις. Μια κυρία είπε ότι δεν θέλει να είναι γυναίκα των ποσοστώσεων ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, ότι οι γυναίκες έχουν τελείως διαφορετικές ε, ανάγκες όσον αφορά την παρουσία τους ε, στις διοικήσεις, ε, αυτό είναι σωστό. Όσον αφορά την τροπολογία 44, έχω καταστήσει σαφές ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την προστασία και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις πράσινες θέσεις εργασίες αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλέ διαφορετικέ επιχειρήσει Εάν μεταφερθεί μέρο τη παραγωγή μα σε χώρε ε, που δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, αυτό θα είναι μια ε, εξέλιξη την οποία ναι, εντάξει μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει, αλλά... Μπορεί κάποιε χώρες οικονομικά να μην είναι σε θέση να προστατεύσουν το περιβάλλον, αλλά πολλές φορέ λείπει και η οικολογική κατανόηση. Γι' αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε στον τομέα αυτόν και θα ήθελα πρέπει να ακούσω τη θέση, ε, τη θέση σου. Ευχαριστώ ε, και για την ε, διάθεσή σου να συνεργαστείς. Συγχαρητήρια για την έκθεση και νομίζω ότι με βάση του συμβιβασμού θα μπορέσουμε να πετύχουμε ευρεία συμφωνία διότι αξίζει τον κόπο στην έκθεση αυτή να πετύχουμε ευρεία στήριξη. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν και μετά η κυρία Πλάμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ισχυώδη συζητητή μα, ο κύριο Στέρξ, δεν είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να κάνω κάποιε παρατηρήσει ε, στο όνομά του. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Μου είπε ο κύριο Στέρξ ότι κατά τη συζήτηση τη έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την ε, σχέση με την ε, στρατηγική 2020 τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά κάποιε τροπολογίε. Η τροπολογία 32. Ο κύριο Στέρξ δεν συμφωνεί με τον αποκλειστικό κατάλογο τομέων δεν, δεν συμφωνεί με τον εξαντλητικό κατάλογο και έτσι αποκλεί κάποιες κάποιους τομείς. Όσον αφορά την τροπολογία 40, ε, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική την Απασχόληση πιστεύει ότι ήδη συμπεριλαμβάνεται στη Στρατηγική 2020 με διάφορους στόχους. Ε, θεωρεί λοιπόν ότι είναι περιττό να δημιουργηθεί νέα στρατηγική, η δεύτερη στρατηγική. Όσον αφορά την τροπολογία 60, συμφωνεί ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και δεν συμφωνεί με την ποσόστοση. Προσωπικά εγώ διαφωνώ μαζί του, διαφωνώ ε, και με την ε, εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Υπάρχει και μια άλλη τροπολογία, νομίζω ότι είναι η 95, ε, μπορεί αυτή να είναι υπερβολικά ευρεία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω με τις ποσοστώσεις. Τροπολογία 61 όσον αφορά τις επισφαλείς θέσεις εργασίας είπε ότι υπάρχει Κίνδυνο σε όλες τις χώρες, για παράδειγμα στο Βέλγιο. Το να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα πλαίσιο ε, για ε, ε, αντιπροσωπευτικούς φορεί, αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση Και τέλος, τροπολογία 79 είπε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, στο Βέλγιο, για παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να ε, θεσπίσουν έναν αντιπροσωπευτικό φορέα. Και τέλος, όσον αφορά τον φόρο του ΜΠΙΝ, ε, δεν μπορεί να συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με κάτι τέτοιο. Αυτές είναι γενικά οι θέσεις του. Συμμερίζομαι πολλές από αυτές, όχι όλες, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να έχουμε διμερείς επαφές με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ τελευταία εισηγήτρια, ε, η τελευταία μιλήτρια στο κατάλογο είναι η κυρία Πλάμ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σρέντερ για το επικοδομητικό διάλογο και το πνεύμα συνεργασίας που επικράτησε στις συνομιλίες μας. Εγώ θα είμαι η συγγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα ήθελα μετά τη συζήτηση που είχαμε να παρακαλέσω την κυρία Σρέντερ να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να ελοπίσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι οικονομικές πολιτικές και κυρίως οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές πολιτικές δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους ούτε σε εθνικό ούτε σε τοπικό αλλά ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι συμπληρωματικές όλες αυτές οι πολιτικές και για να επιτύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Γι' αυτό και καλό θα είναι να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να χρησιμοποιήσουμε τους καλύτερους τρόπους και να μιμηθούμε τις βέλτιστες πρακτικές για να ε, επιτύχουμε ένα υφόρο μοντέλο εργασίας. Ας μην ξεχνούμε και τον ορισμό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τον ορισμό για τις πράσινες ε, θέσεις εργασίας που θα είναι και αξιοπρεπείς, θα εξασφαλίσουν και μια σωστή μετάβαση προς μια βιώσιμη και υφόρο οικονομία. Σας ευχαριστώ κύριε Σρέντερ και παρακαλώ μην ξεχνάτε τις παρατηρήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ε, η κυρία Φιγκερέδο μπήκε τελευταία στον κατάλογο των ομιλητών, αλλά άλλο δεν θα δεχτώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή μας, κάτι που ήδη είχα πει στην εισηγητρία, ότι είμαι η συντάκτρια γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας για την έκθεση της κυρίας Σρέντερ. Η γνωμοδότηση, μάλιστα, θα ψηφιστεί σήμερα την ίδια ώρα που θα ψηφίζουμε εμείς την έκθεση για το ελάχιστο εισόδημα. Γι' αυτό και θα απουσιάσω στην ε, ψηφοφορία αυτή, γιατί επαναλαμβάνω συμπίπτει με την ψηφοφορία της δικής μου γνωμοδότησης στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Πάντως ε, και η γνωμοδότηση περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις και ελπίζω να τις λάβει υπόψη η συγγήτρια στην τελική διαμόρφωση της έκθεσής της. Ευχαριστώ. Ε, Εισηγητή, για να Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους. Έχω σημειώσει επιμελώς τα όσα μου είπατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται πιο σύντομα. Πρώτα, το θέμα των μελετών για τις μελέτες έκανα την επιλογή μέσα στην έκθεση να βασιστώ στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτά δηλαδή που χρησιμοποίησε για την έκθεσή της employment, ε, χωρίς να ε, εξετάσω άλλες μελέτες. Παρόλο που εγώ βέβαια διάβασα πολύ περισσότερες. Και βέβαια θα ήταν ανεξάρτητος ο κατάλογος εάν δεν περιοριστώ σε αυτά. Δεύτερο, Σάρι Σάια. Ναι, αν πρέπει να ενταχθεί στο σύνολο της οικονομίας, ναι. Και έχουμε περιλάβει και πολλές από τις προτάσεις σας σε συμβιβαστικέ τροπολογίες. Θα τα δείτε αυτά. Περιέλαβα και αυτό που είπατε, ότι δηλαδή υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις ό,τι αφορά τιμολόγια, κοινωνικέ εταιρικέ σχέσει κλπ. στι διάφορε χώρε μέλη. Πάλι εγώ έχω κάνει σχετική τροποποίηση σύμφωνα με τι προτάσει σα. Αλλά έλαβα και προτάσεις που έλεγαν ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να το έχει κανείς υπόψη του και αυτό. Έλεγαν για παράδειγμα για ορισμένες χώρες μέλη, γι' αυτό το λέμε δηλαδή τελικά στην, ε, στην ε, συμβαστική τροπολογία για ορισμένες χώρες μέλη ή πάντως λέμε όχι για όλες τις χώρες μέλη. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Τώρα υπόθεση των ποσοστώσεων. δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο γιατί έχει υποβάλει μια σχετική πρόταση και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Εγώ πάντως δεν θα επιμείνω στην δική μου διατύπωση. Θα φροντίσω να γίνει ψηφοφορία για τις τροπολογίες της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών. Έξτρα αυτό, επειδή κατανοώ ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, θέσεις, υπάρχουν από την άλλη μεριά ακριβώς αντίθετες θέσεις. Η Επιτροπή Γυναικών έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω πάντω ότι η δική μου διατύπωση είναι... Η διατύπωσή τους είναι καλύτερη, γι' αυτό και εγώ παρετούμε από τη δική μου. Ας γίνει λοιπόν η ψηφοφορία και θα δούμε που θα καταλήξει και έτσι δίνουμε και το δικαίωμα στην ε, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών να ε, ψηφιστούν οι τροπολογίες της. Βέβαια εμείς διατηρούμε την αρμοδιότητα επί της ουσίας. Τώρα και για τις Γνωμοδοτήσει της Επιτροπής Περιβάλλοντος και άλλων προσπαθήσαμε να τις περιλάβουμε όλες και να τις βάλουμε στις ε, σωστές θέσεις μέσα στην έκθεση. Ορισμένες βέβαια φύγουν τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής, οπότε η δική μας ε, Επιτροπή θα επιμείνει σε αυτά που θεωρεί ότι είναι ε, της δικής της αρμοδιότητας και είναι και πιο συγκεκριμένα. Αλλά όπου αρμοδιότητες ανήκουν σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, τα πράγματα μένουν έτσι, θα έρθουν στην ψηφοφορία διατηρούνται και εντάσσονται στα οικία μέρη. Το ίδιο και για την Ήλντα. Περιμένουμε ακόμα. Η Ήτρε θα κάνει πολλά για τις συνθήκες πλαίσια, όπως έκανε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ένβη, και θα τα δούμε και θα τα ψηφίσουμε. Διατηρούνται όμως, θα είναι και μακρύς ο κατάλογος των ψηφοφοριών, πάντως θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα. Τώρα για την βιώσιμη ή πράσινη είναι δύσκολη η υπόθεση αυτή. Εμείς προσπαθήσαμε πάντως να περιλάβουμε την πρόταση αυτή. Κατάλαβα τι εννοείται ότι θέλετε να έχουμε την ίδια διατύπωση. Από την άλλη μεριά, από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές μας δίνουν άλλα, άλλες προτάσεις που έχουν την ορολογία πράσινη μέσα. Πάντως ε, πολλές από αυτές τις περιλάβαμε κυρία Σάιερ. Για τον κύριο Στέρξ, για την ε, πολιτική 2020 έχουμε κάνει εντονότερες τις διασυνδέσεις. Θα μπορούσα να μιλήσω μαζί σας, αλλά δεν μπόρεσα. Προσπάθησα πολλές φορές να μιλήσω μαζί του, αλλά δεν τα κατάφερα. Η κριτική δεν είναι ότι περιλαμβάνεται στην Ευρώπη του 2020, εμείς τα ενισχύσαμε τα σημεία αυτά. Η κριτική είναι ότι δεν εμφανίζουμε αυτά τα αποτελέσματα των συνεργειών, τα οποία εμείς τα συζητήσαμε και με την Βελγική Προεδρία, η οποία είναι διατεθειμένη να βελτιώσει το σχετικό κείμενο. Και αυτές τα αποτελέσματα των συνεργειών θα βελτιωθούν. Θέλει να το αναλάβει αυτό η Βελγική Προεδρία. Θα δούμε λοιπόν τώρα πώ μπορούμε, πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες διατυπώσεις που να μην δείχνουν ότι είμαστε κατά της ε, πολιτικής 2020, της του 2020, αλλά ότι θέλουμε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των συνεργειών. Ελπίζω να καταφέρω να συναντηθώ μαζί του κάποια στιγμή και να μιλήσω μαζί του. Τώρα, για τι κοινωνικέ εταιρικέ σχέσει, εγώ θα επανεξετάσω, αν θα ενταχθεί δηλαδή στι χώρε μέλη, θα επανεξετάσω τώρα την διατύπωση για, τις, ε, για τους ορισμούς της ε, Οργάνωσης Εργασίας. Εγώ ε, για τις ε, πράσινες εργα... Ε, θέσεις απασχόλησης θα δεχθώ αυτά που λέει ο κύριος Μαν. Δικές του είναι βασικά οι τροπολογίες, άλλωστε το δέχτηκα εγώ αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει ιδεοδό να συμφωνήσουμε όλοι στο ίδιο κείμενο το δικό του. Και για τη δική του τροπολογία 44 βέβαια την δέχομαι, πρόκειται για μια προσθήκη και ασφαλώς την δέχομαι χωρίς κανένα πρόβλημα. Άλλωστε δεν υπάρχει και κανένας ανταγωνισμός σε αυτήν την ε, ε τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Σρέντερ στη συνεδρίαση της 13ης και 14ης Ιουλίου. Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας και λείπουμε για την πεντάλεπτη καθυστέρηση. Ελπίζω να έχετε όλοι μαζί στις ηλεκτρονικές κάρτες, αν θα ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση Μωρά, γνωμοδότηση για την ακρίβεια, με θέμα τη χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Για την παράγραφο 1 ψηφίζουμε την τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Μάλλον έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Κύριε Κύριε Κρίστινσεν, ξεχάσατε την κάρτα σας. Τι ψηφίζετε. Υπέρ. Ωραία. Euh, Ξέχασε κανείς άλλος την κάρτα του. Ψηφίζετε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εσείς τι ψηφίζετε κατά. Ούτως ή άλλως 15 υπέρ, 22 κατά. Έχει σαφώς απορριφθεί. Τροπολογία 4 με ρόιτε ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγράφω. 1, τροπολογία προφορική. Θέλετε να μας την παρουσιάσετε κυρία Μωρά. Βεβαίως. Υποβάλλουμε προφορική τροπολογία για την οποία υπάρχει συμφωνία ώστε να συνδυάσουμε την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με το Ταμείο Συνοχής και λέμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την συνέχιση του EGF και την αναμενόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση του Κοινωνικού Ταμείου στην αναθεωρημένη εκδοχή του 2009 Θέλουμε να μπορούμε να αντιδράσουμε σε κατεπίγουσες περιπτώσεις ε, και σε καταστάσεις κρίσης. Αυτή την προφορική τροπολογία θέλω να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με τέσσερις ψήφους κατά. Τροπολογία 5. Κορνέλισεν για την παράγραφο 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Τώρα μετά την παράγραφο 2, τροπολογία 9 της κυρίας Χάρκιν και τους συζητητές των τριοδομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2 έχουμε τη συμβαστική τροπολογία α. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 τώρα. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 συμβατή. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 κατά καταπίπτει. Μετά την παραγραφό 3, τροπολογία 14 πολλών συντακτών. που είναι υπέρ, κατά αποχές. Τώρα, μετά την παραγραφό 3, 15, θα ψηφίσουμε την τροπολογία χωρίς το προετοιμάζοντας την εφαρμογή. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 15, με εξαίρεση αυτή τη φράση, κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της προσθήκης αυτής της φράσης, κατά αποχές Όχι, κατέπεσαν αυτές οι λέξεις. Μετά την παραγραφό 3, τροπολογία 16 τη κυρία Κορνέλη είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 17, Χέντελ υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 18 του ιδίου, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 19 του ιδίου υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 20 του ίδιου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 τροπολογία Νταρντέν ποιος είναι υπέρ για την 4 κατά αποχές εγκρίνεται 22 της κυρίας Ρόιτ είναι συμβατή ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά την παράγραφο 5 23 πολλών συντακτών ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 24 ε, Κορνέλισεν μετά την παράγραφο 5. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 τροπολογή 25. Γκρούνι και Μωράν Σαρτιέ, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 26, Κορνέλης υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάλι για την παραγραφή 6, τροπολογία 28, είναι γλωσσική. Euh, γλωσσική τροπολογία αφορά την αγγλική μετάφραση. Κυρία Πρόεδρε, η Μαρία Χάρκιν πέσει την προσοχή μας στο γεγονός ότι ήταν ασυνάρτητη η αγγλική μετάφραση στο σημείο αυτό και γι' αυτό προτείναμε τη γλωσσική τροπολογία για να είναι πιο εύληπτη η φράση αυτή. Δεν θα ψηφίσουμε τη γλωσσική τροπολογία. Τι ουσιαστικέ τροπολογίε ψηφίζουμε. Οι γλωσσικέ τροπολογίε δεν τι ψηφίζουμε κανονικά. Κυρία Πρόεδρε, όμως επιτρέπετε, ο τύπο έχει σχέση με την ουσία, η διατύπωση έχει σχέση με την ουσία, γι' αυτό θα πρότεινα να ψηφίσουμε και αυτή την τροπολογία και τη γλωσσική. Το γαλλικό κείμενο λέει καλεί τα κράτη-μέλη που αποφελούνται ε, από το ταμείο αυτό να είναι πιο ελαστικά και να ε, με μεμονωμένη προσέγγιση εξατομικευμένη για τους απολυμμένους εργαζομένους. Το αγγλικό κείμενο λέει καλεί τα κράτη-μέλη είναι αποτελεσματικά και να υιοθετήσουν προσωπική προσέγγιση. Και η τροπολογία της ηγήτριας προτείνει να βελτιώσουν την ε, αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και να υιοθετήσουν εξατομικευμένη προσέγγιση. Αυτό λέει η γλωσσική τροπολογία 28. Αν όμως ε, εγκρίνουμε αυτή την γλωσσική τροπολογία θα πρέπει να τροποποιήσουμε και το γαλλικό κείμενο. Γιατί αν πούμε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής θα πρέπει να αλλάξουμε και την γαλλική μετάφραση, γιατί είναι τελικά ουσιαστική, δεν είναι καθόλου μόνο απλά γλωσσική. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη, δηλαδή και στη γαλλική μετάφραση, να πούμε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα εφαρμογή του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση. Άρα είναι ουσιαστικότατη τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 28, όπω έχει τροποποιηθεί. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 είναι συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 συμβατή και αυτή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την παράγραφο 7 συμβαστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 καταπίπτει καθώς και οι ακόλουθες. Μετά την παραγραφο 7 έχουμε την τροπολογία 37 της κυρίας Χίρς, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 7 έχουμε την τροπολογία 38. Κορνέλησεν. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 39. Όμπερμαϊρ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 40. Το 2. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Για την παράγραφο 8. 41 Τη κυρία Κορνέλης υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 17 ψήφισαν υπέρ, 20... 16 ψήφισαν υπέρ, 23 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. 43 ο Μπερμάιρ. 42 μάλλον ο Μπερμάιρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 43. Στάινρουκ. Συμβατή. Ποιο είναι υπέρ τη 43. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44. Του κύριο Ντάρντεν. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 πολλών συντακτών. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 για την παραγραφή 9. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9, τροπολογία 47, έχει καταπέσει όμως γιατί καλύφθηκε από τη συμβαστική λύση. 48, Κορνέλησεν, ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε μέχρι τα ταμεία. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παραγραφή 9, 49 πολλών συντακτών, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 50 της κυρίας Πλάμπ, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 52 της κυρίας Κορνέλησεν, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54, παραγραφό 11. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 11, τροπολογία 55 του κυρίου Χέντελ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την 11 παράγραφο, τροπολογία 56 της κυρίας Χίρς, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12, 55, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές 53 συγγνώμη του κύριου Χέντελ αποχές εγκρίνεται 57 του κύριου Ντέρντεν καταπίπτει το ίδιο και 58 Αιτιολογική σκέψη τώρα, αιτιολογική σκέψη α, μετά την αιτιολογική α, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη β, τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι τέλος. 33 ψήφοι υπέρ. Μία ψήφος κατά. 34 μάλλον ψήφοι υπέρ. Μία ψήφος κατά και 7 αποχές. Θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Nous en venons euh, au point 10, au vote du... Σημείο 10 τώρα, ψηφοφορία της έκθεσης Φιγκερέντο. Με θέμα το ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία Ι. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες καταπίπτουν. Μετά την παραγραφό 1, τροπολογία 70 της κυρίας Ροντζούλη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 της κυρίας Δελή, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 72, Γκέντς και Στάινρουκ, ποιος είναι υπέρ, με προφορική τροπολογία που λέει... Επισήμαστε την πρόεδρο να μιλάει λίγο πιο αργά. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 72 των κυρίων Γκέντς των κυριών Γκέντς και Στάινρουκ. Έχουμε και προφορική τροπολογία που προσθέτει μετά το αντιμετωπίζει ότι. Προσθέτουμε one-off. Μία από τις πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους. Ποιος είναι υπέρ της 72 με προφορική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 μετά την παραγραφή 1 του κ. Πουπάκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 Ποιο Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 της κυρίας Ροντζούλη. Με προφορική τροπολογία της κυρίας Φιγκερέντο. Και πάλι προσθέτει ένας από τους πιο one-off, πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 του κύριου Πουπάκη Αργά μιλάω, πιο αργά δεν γίνεται, λέει η πρόεδρος. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 76 του κυρίου Πουπάκη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 77 του κυρίου Πουπάκη. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Συμβαστική τροπολογία J από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2. Τροπολογία 86 της κυρίας Κρέτσου. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικό έλεγχο αν και μάλλον έχει απορριφθεί, για την τροπολογία 85, τη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 19 υπέρ, 22 κατά. Όντως απορρίπτεται. 88, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, τροπολογία 89 του κ. Νταρντέν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 της κυρίας Φιγκερέντο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 91. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Δίκιο έχετε κυρία Φιγκερέντο. 23 ψήφοι υπέρ, 19 κατά και μία αποχή, άρα εγκρίνεται η τροπολογία 91. Τροπολογία 92 τώρα, γλωσσική τροπολογία και άρα δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 93. το κύριο Νταρντέμ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ο λάθος, λάθος, λάθος, απορρίπτεται. Ή Μάρα, να το επαληθεύσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. 93. Ψηφίσατε όλοι. ψηφοφορίες. ψηφοφορίας. 22-22 ισοπαλία, άρα απορρίπτεται. 94 Φιγκερέντο, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Με ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα μέχρι μέσω κινήτρων. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος της 96. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε δεν έχει νόημα το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 97 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία συμβαστική κάπα στην παράγραφο 3 από τρεις ομάδες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε οι σχετικές τροπολογίες καταπίπτουν. Παράγραφος 3. Τροπολογία 110 έχει καταπέσει όμως, ε, επειδή υιοθετήσαμε την συμβαστική τροπολογία Κ. Θα ψηφίσουμε την παράγραφο 3. Όχι, διορθώνει η πρόεδρος. Η παράγραφος 3 Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί, γιατί εθετήσαμε τη συμβαστική τροπολογία Κ, μετά την παράγραφο 3. Τροπολογία 111 της κυρίας Ραντζούλη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 112 του κρυπού Πουπάκη Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113. Όμπερμαερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114. Νταρντέν. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 δελή υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας 19 ψήφισαν υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. Μετά την παραγραφό 3, τροπολογία 116 της κυρίας Γκρουνή, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα μέχρι εκτός της φτώχειας, να βγουν από τη φτώχεια. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται, το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. 117 αντελεί ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 119 γκρούνι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 120 ροντζούλι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 121 της κυρίας Δελή υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Για την παράγραφο 4 έχουμε τη συμβαστική τροπολογία L από τέσσερις ομάδες που είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, 128 της κυρίας Φιγκερέιδο, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 129 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 131 της κυρίας Τσίμερ και του κυρίου Χέντελ. Με προφορική τροπολογία της κυρίας Ντελή που λέει σύμφωνα με την γραπτή διακήρυξη παριθμών 111 του 2007. Και επίσης προσθέθηκε μια νέα παράγραφο ανάγκη να μετατραπούν οι κατευθυντήρες γραμμές για τη φτώχεια σε συγκεκριμένους εθνικούς και υλοποιήσιμους στόχους για θέματα προτεραιότητες για την κοινωνική στρατηγική που δεν αποκλεί κανέναν. Ωραία, αφού δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε την 131, την αρχική, χωρίς την προφορική τροπολογία της κυρίας Δελή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, αν και πιστεύω ότι έχει απορριφθεί η τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 19 ψήφισαν υπέρ, 25 κατά. Μία αποχή, άρα φως φανάρι απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 130 της κυρίας Δελή. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν της κυρίας Γκρούνη. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Ηλεκτρονικός έλεγχος, Άρχιτε ψηφοφορία. Μου να πει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 8 κατά και 14 αποχές. Εγκρίνεται. 133 της κυρίας Δελή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. 134. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της 134. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135 Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 134. Αλλά θα δείτε ότι δεν έκανα λάθο ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε όλοι, τέλο. 21 υπέρ, 23 κατά. Δεν ήταν τόσο σαφές βέβαια το αποτέλεσμα, αλλά παρόλα αυτά απορρίπτεται. 135 των ιδίων της κυρίας Τσίμερ και του κυρίου Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Ε, καλά, λάθος έκανα. Παράγραφος 5. Συμβαστική τροπολογία M. Μη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται σαφέστατα. Μετά την παραγραφό 5 έχουμε την 138 της κυρίας Φιγκερέντο υπέρ κατά εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 5 149 της κυρίας με προφορική τροπολογία της κυρίας Φιγκερέντο Υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία καταρχήν. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την 149 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 5, 120 τροπολογία Σκύρια Τσίπερ. 150 μάλλον, 120 λέει η 150, ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπάρχει ένα λάθος στους καταλόγους ψηφοφορίας. 152 τροπολογία δεν έχει αποσύρθει. 154 είναι που αποσύρθηκε. Οπότε ψηφίζουμε την 152 Φιγκερέντο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται η 152. 153 της κυρίας Ντελή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 153. Tout le monde le vote όλοι τέλος. Ψήφισαν 21 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Η 154 έχει αποσυρθεί. 155 της κυρίας Ντελή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 155. 156 του κύριου Πουπάκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 του ίδιου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 158 της κυρίας Ντελή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. 159 αντελεί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή για την παράγραφο 6. Συμβαστική τροπολογία νη. Τεσσάρων ομάδα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6. Τροπολογία 165 της ηγετρής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παραγραφή 6, τροπολογία 167 του κυρίου Νταρντέν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 της κυρίας Γιαρόκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 170 Ποιο είναι υπέρ τη κυρία Φιγκερέτο κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την παράγραφο 7 συμβαστική τροπολογία ο μικρόν. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 7 179 τη κύρια Ροντζούλη ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181, το κύριο Πουπάκη, με προφορική τροπολογία του. Διαγράφει το on an equal footing. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ποιος είναι υπέρ της 181. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 πουπάκι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 183 του ίδιου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 184 ροντζούλι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. «185» της κυρίας Κρέτσου Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφή 8, τροπολογία 186, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 186. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. όλοι. Τέλος. 34 υπέρ, 11 κατά. Δίκιο έχετε κυρία Μαν. Εγκρίνεται 186. 187 τώρα με προφορική τροπολογία της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ της 187? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θεωρώντας τώρα, το μετά το πρώτο θεωρώντας, τροπολογία 1, τριών συντακτών, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θεωρώντας 2, τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το θεωρώντας 5, τροπολογία 6, με προφορική τροπολογία της ηγήτριας. Αντιρρήσεις δεν υπάρχουν, ψηφίζουμε την τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α γιατί τη θεωρώντας 16, πιο είναι κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το θεωρώντας 16, τροπολογία 10 της κυρίας Ντελή. ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το 17, τροπολογία 11, κυρίων Γκέντς και Σάινμπρουκ, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα, μετά την α, τροπολογία 12, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το β, συμβαστική τροπολογία β, τεσσάρων ομάδων. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την ιτηλογική σκέψη Β, τροπολογία 15, ποιο είναι υπέρ, της Δέλη, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16, Γκέντ και Στάινρουκ, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το Δέλτα, 17 τροπολογία, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για τα ε 18 τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 της κυρίας Ροντσούλη, Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σε από τέσσερις ομάδες, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το F τροπολογία 23, των κυρίων Τσίμερ Φιγκερέντο και του κυρίου Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη F, τροπολογία 24... Τσίμερ, Φιγκερέδο και Χέντελ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά το απολογή 25 της κυρίας Ντελή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 28 υπέρ, 16 κατά. Μία αποχή. Όχι λάθος λέει πρόεδρος. 27 υπέρ, 17 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται η τροπολογία 25. Τροπολογία 26 της κυρίας Ντελή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάλι της κυρίας Ντελή, τροπολογία 22, ποιος είναι υπέρ, κατά, οχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Κώστα και Καετάνο. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F για την αιτιολογική σκέψη K. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 κύρια Ροντζούλη υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά το L, συμβαστική τροπολογία G, τεσσάρων ομάδων, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H, τεσσάρων ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την ιδεολογική σκέψη M, τροπολογία 52, τον κυρίων Κοφεράτη, Κώστα και Μπαλτασάρ. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 της κυρίας Κρέτσου, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 Κρέτσου, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. 56 Φιγκερέντο, ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. 57 της ηγετρίας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 της ίδιας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε, Κλωσική. Και τροπολογία 20 της ηγετρίας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε Α, συγγνώμη, κύριος Νταρντέν. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα με δύο λόγια να εξηγήσω την ψήφο που θα δώσουμε στην έκθεση. Θα απόσχουμε τελικά. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε την έγκριση έκθεσης, γιατί συνιστά πρόοδο και είδατε ότι δείξαμε θετική στάση για πολλές συμβαστικές τροπολογίες, ιδιαίτερα τη συμβαστική τροπολογία M, αλλά διαπιστώνουμε ότι οι παράγραφοι της γνωμοδότησης, της έκθεσης, έχουν απορριφθεί με οριακή ψηφοφορία, αλλά παρόλα αυτά απορρίφθηκαν. Έχουμε την αίσθηση ότι μέχρι την Ολομέλεια θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο, γι' αυτό και θα κρατήσουμε στάση αποχή ως ομάδα. Ευχαριστώ. Κυρία Φιγκερέντο. Δεν θα επανέλθουμε τώρα στη χθεσινή συζήτηση. Αυτή έγινε. Ήθελα να κάνω μόνο δύο σύντομες παρατηρήσεις. Λυπούμε ειλικρινά που δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρώσουμε μία πλειοψηφία υπέρ της οδηγίας. Έδωσα μάχη μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά όπως φάνηκε και σήμερα δεν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πλειοψηφία υπέρ της οδηγίας, υπέρ της έκθεσης. Δεύτερον, παρά αυτή την ανεπάρκεια και τις αδυναμίες της έκθεσης, πιστεύω παρόλα αυτά ότι έχει κάποιες θετικές προτάσεις, μία δειλή πρόοδο που δίνουν κάποια σημάδια, κάποια μηνύματα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να δείξουν μεγαλύτερη προσήλωση στην ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας στο έτος αυτό που έχουμε. Τη καταπολέμηση τη φτώχεια. Και θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προ σοσιαλιστές να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τον Οκτώβριο να υιοθετήσουμε μια έκθεση που θα είναι βελτιωμένη, μια βελτιωμένη εκδοχή τη ε, της σημερινής. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ψηφίσω υπέρ. Άλλο κανεί θέλει να εξηγήσει την ψήφο του, τη στάση του πριν την τελική ψηφοφορία. Mm. Κυρία Ορή, όχι. Οπότε άρχεται η ψηφοφορία τελική για την έκθεση Φιγκερέντο. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 23 ψήφισαν υπέρ, 5 κατά και 14 αποχές. Η έκθεση εγκρίνεται. Ευχαριστούμε θερμά την εισηγητριά μας για τις προσπάθειες που κατέβαλε να συντάξει συμβαστικές λύσεις και να βρει συμφωνία. Nous en venons ακολουθεί το 11 όπου ησυχία παρακαλώ όπου θα εξε, εξετάσουμε τις τροπολογίες και τις κατήφθες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών. Τον λόγο θα λάβει ο εισηγητής κ. Ορή. Merci bien, madame. Euh, Α, θα μιλήσω καλύτερα ουγγρικά, λέει ο κύριο Σωρή. Euh, Η Πρόεδρος, σας παρακαλώ, δείξτε σεβασμό σε όσους επιθυμούν να εργαστούν. Παρακαλώ, αποχωρήστε με ησυχία. Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καμιά φορά τα πράγματα στη διάρκεια της σύνταξης της έκθεσης ήταν εύκολα, καμιά φορά ήταν δύσκολα. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους ε, για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για την έκθεσή μου. Βλέπετε κατέθεσαν 294 τροπολογίες, από από συνολικά 34 βουλευτές. Δηλαδή σχεδόν όλοι οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής θέλησαν να κάνουν κάποιες προτάσεις. Παρά τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών, η πλειοψηφία τους είναι τέτοια που μπορούν να ενταχθούν με κάποιο τρόπο στο κείμενο, ώστε το κείμενο πραγματικά δεν διαλύεται λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των τροπολογιών. Νομίζω μάλιστα ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες και αυτό θα οδηγεί σε σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού τους. Και εν τέλει το κείμενο νομίζω θα είναι ε, εύκολο να γίνει αποδεκτό. Πάντως όπως είπα ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους τους συναδέλφους. Βέβαια υπάρχουν και δυσκολίες. Ο αρχικός στόχος μου ή ας πω καλύτερα η αρχική μου πρόθεση ήταν να καταλήξουμε ίσως σε 15-20 συμβαστικές τροπολογίες σε θέση των περίπου 300. Ελπίζω, ελπίζω να μπορέσω να τηρήσω περίπου αυτόν τον στόχο. Εκτός του προημίου τώρα και της κατευθυντήρας γραμμής 10, όπου και εγώ ίδιος κατέθεσα τροπολογίες επί του αρχικού κειμένου, δηλαδή αν εξετάσετε το αρχικό κείμενο της ε, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εννοώ, εγώ επιζητώ κάποια αναπροσαρμογή του, μπορούμε να δούμε ποιε τροπολογίε θα δεχτούμε και ποιε όχι και μετά να ψηφίσουμε, αλλά σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες 7 και 8, αλλά και την 9, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ε, επιλύσουμε είναι ποιο κείμενο για αυτές θα λάβουμε ως βάση. Το κείμενο της Κομισιόν θα το λάβουμε αυτό ως βάση ή θα λάβουμε ως βάση την δική μου πρόταση που θα οδηγήσει σε νέα δομή. Και τότε θα πρέπει να συγχωνευτούν οι αρχικές κατευθυντήριες γραμμές 8 και 9 όπου μιλούμε για τα σχολικά συστήματα, για την εκπαίδευση εκτός σχολικών συστημάτων και άλλα σχετικά θέματα. Εγώ έχω συλλέξει ορισμένες σχετικές πληροφορίες. Τα οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές σε αυτά αναφέρονται. Πρέπει επίσης να δούμε τη σημασία του να επιτεθούν οι στόχοι της απασχόλησης δια της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Ε, εγώ νομίζω ότι σε αυτές πρέπει να εμείνουμε στο κείμενο. Και οι τροπολογίες εκείνες που αναφέρονται στις κατευθυντήρες γραμμές 7, 8 και 9 είναι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί επί του αρχικού κειμένου της Κομισιόν. <clears throat> Ας δούμε λοιπόν κατά πόσον μπορούν να ενταχθούν χωρίς καμία δυσκολία στο νέο κείμενο. <clears throat> Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν ο πρώτος προβληματισμός που αντιμετώπισα. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εδώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Έχουμε ήδη κάνει δύο σχετικές συζητήσεις. Έχω καταθέσει και εγώ ορισμένες τροπολογίες με στόχο να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους συναδέλφους στις προηγούμενες συζητήσεις. Άρα υπάρχει και σε κάποιο βαθμό μια επανάληψη και κάποια σύγκληση πάλι μέσα στα πλαίσια της αναζήτησης κάποιων συμβιβασμών. Μιλούμε για απασχόληση ποιότητας, για απασχόληση αξιοπρεπή ε, στον τίτλο αυτό και έχουμε εδώ ορισμένα σχόλια που έγιναν από συναδέλφους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αλλά και από άλλες ομάδες και εγώ κατέθεσα μια τροπολογία σχετικά με το concept, αλλά μπορούμε να κάνουμε το κείμενο λίγο πιο ακριβές, ώστε εν τέλει να μπορέσει να ενταχθεί ε, στην έκθεση. Και επίσης οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτε έχουν κάνει ορισμένε τροπολογίε σχετικά με τον απότερο στόχο που είναι η πλήρης απασχόληση. και μιλούμε για αυτές τις καθηγητές ότι θα διαρκέσουν για μια δεκαετία. Μπορούμε να το περιλάβουμε αυτό στο κείμενο. Όλα τα βασικά κείμενα της Ένωσης, αλλά και, ό, και όσα λένε τα διάφορα πολιτικά κόμματα, όλοι έχουν αναλάβει δέσμευση για να καταπάνουν προσπάθειες για τη δημιουργία πλήρους απασχόλησης. Άρα μπορούμε να το εντάξουμε στο κείμενο. Βέβαια, επιλέγοντας μια διατύπωση που να είναι κοινά αποδεκτή. Επίσης, ε, γίνεται λόγος για πιο αποτελεσματικό monitoring, το οποίο εμένα επίσης με απασχολεί πολύ. Βρήκα ορισμένες έξοχες ιδέες ανάμεσα στις τροπολογίες που μου υποβλήθηκαν. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε μέσω μιας συμβαστικής τροπολογίας σε ένα πραγματικά πολύ καλό κείμενο. Το ίδιο ισχύει και για το εξής. Ορισμένοι υποστηρίζουν και εγώ με δική μου τροπολογία επίσης για την πρόσβαση των νέων δηλαδή στην αγορά εργασίας ως ιδιαίτερο στόχο, ως ένα είδος υπό στόχο. Πολλοί μου μίλησαν γι' αυτό. Όταν μιλούμε δηλαδή για μια απασχόληση της τάξης του 75%, μιλούμε πάλι για ορισμένες ομάδες ηλικιών και η ομάδα ηλικίας 15-24 ετών πρέπει να ε, συζητηθεί εδώ. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ε, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία ή θα πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος, αλλά όπως είπα υπάρχουν ορισμένες διαφορές. Υπάρχει πάλι διαφορά αν μιλούμε για τα, τους νέους που είναι 20-24 ετών. Ε, και όχι 15-24 ετών. Και σε ό,τι αφορά άλλε ηλικιακέ ομάδε, 24 έω 64 ετών, εκεί χρειάζεται να το δούμε ξανά. Εγώ θα υποστηρίξω τις προσπάθειες αυτές βέβαια. Θα υποστηρίξω τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί σε αυτές τις ε, τροπολογίες, αλλά όπως είπα πρέπει το κείμενο να γίνει ακόμα πιο λεπτομερές και ακριβές. Για να προσφερθεί για παράδειγμα ε, μια προστασία, μια υποστήριξη σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν ε, από την ε, απαραίτητη εκπαίδευση. Για παράδειγμα οι ομάδες Ρωμά. Το ίδιο σημαντική είναι μια κοινωνική οικονομία και βέβαια εν ώψη της κρίσης που ζούμε. Έχουν εγερθεί και φωνές κριτικής σχετικά με το ότι έχουμε αφήσει εκτός την απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Βλέπω και εγώ ότι υπάρχει δίκιο στην άποψη ότι πρέπει να ενταχθεί και αυτή η απασχόληση. Το μιλούμε δηλαδή σε ορισμένε τροπολογίε για αυτού που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα. Θα δεχτώ λοιπόν και αυτή την επιθυμία. Και όπως είπα, η απόκτηση γνώσεων μέσω της εκπαίδευσης έχουμε την επίσημη, έχουμε και την ανεπίσημη εκπαίδευση και θέλουμε να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ τους και να τους δοθεί η ισότιμη βαρύτητα μέσα στο κείμενο. Εγώ θα το υποστηρίξω αυτό. Υποστηρίζω και κάποιες πρωτοβουλίες που μιλούν για ένα 10% ε, των προσώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο. Νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε όσο δυνατόν περισσότερους ε, ανθρώπους με προσόντα και όσο το δυνατόν λιγότερους χωρίς. Άρα θα κάνω κάθε προσπάθεια ώστε να μειωθεί το ποσοστό των ε, νέων που αφήνουν το σχολείο. η πολιτική απασχόληση δεν είναι υποσύνολο της πολιτικής συνοχής. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την πολιτική απασχόληση. Αυτό είναι ε, βέβαιο. Όλοι θα συμφωνήσουν. Και εδώ πάλι έχουν γίνει εξαιρετικές ε, προτάσεις και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να τις περιλάβω στο κείμενο. Όπως είπα λοιπόν, νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές που ανέφερα εντάσσονται εύκολα στο κείμενο. Μιλούμε για εσωτερικές και εξωτερικές στρατηγικές και αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Μάλιστα μετά την ακρόαση, τη χθεσινή ακρόαση που ακούσαμε πολλά από τον κύριο Μόντι ήταν εξαιρετική η συνεισφορά του. Και αυτά λοιπόν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε. Και επίσης υποστηρίζω τις προτάσεις εκείνες που λένε ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις αναλογίες. Όπως είπα, εν τέλει αυτή η υπόθεση είναι εθνικής αρμοδιότητας. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας αυτά όταν κάνουμε τις προτάσεις μας και να μην το λησμονούμε. Γίνονται και διάφορες προτάσεις εδώ σχετικά με ε, την ισότητα ανδρών και γυναικών, τα υποστηρίζω και εγώ αυτά με κάποιο τρόπο θα τα συμπεριλάβω στο κείμενο. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθώ με τους κοιόδης σε μια προσπάθεια να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με το πώς μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία στο κείμενο. Έχω ένα πρόβλημα βέβαια με τις προτάσεις των πρασίνων. Όχι όμως πρόβλημα αρχής, γιατί συμφωνώ μαζί τους. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ανάγκη να βάλουμε σε κάθε ε, δεύτερη και κάθε τρίτη παράγραφο την αηφόρο ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικούς συμβιβασμού και για αυτό το θέμα. Βέβαια, ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει περάσει η κρίση, ακόμα δεν βλέπουμε καν φως στο βάθος του τούνελ, αλλά δεν θα ήθελα και να ε, μιλήσουμε μοναχά για τα αρνητικά στοιχεία, να έχουμε ένα είδος δηλαδή αρνητικές αυτοεπαληθευόμενες προφητείες, ας το πω έτσι. Ε, νομίζω ότι η στατική της Λισαβόνας είναι πιο περίπλοκη από τόσο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που θέλουμε ακόμα να κάνουμε στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, αλλά δεν θα πρέπει να μειώσουμε τις προσπάθειες που έγιναν την τελευταία δεκαετία. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου για αυτό. Και μιλώντας εν τέλει για τα κοινωνικά συστήματα, για τις συντάξεις, για την μεταφορά των συνταξιοδοτικών και άλλων δικαιωμάτων μέσα στην ενιαία αγορά. Αυτά έχουν σχέση βέβαια με την κινητικότητα και οι συνάδελφοί μου έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Θα συμφωνήσω, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάλι μαζί τους σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Αυτές οι 294 τροπολογίες φαίνονται εκ πρώτης όψεως σαν ένας τεράστιος αριθμός, αλλά όπως είπα υπάρχουν πολλές τροπολογίες που συγκλίνουν Είμαι λοιπόν αισιόδοξο σχετικά με το τι μπορούμε να επιτύχουμε όταν θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα με τους συναδέλφους μου και οδησίγητες για να καταλήξουμε σε κάποια ενιαία κείμενα συμβαστικών τροπολογιών. Θα διεξέλθουμε και τις 294 τροπολογίες, να δούμε ποιες μπορούμε να δεχθούμε. Κάποιες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν ευθέως στο κείμενο και άλλες όπου θα χρειαστεί περισσότερη μελέτη. Πάντως Ξαναλέω ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθώ με του συναδέλφους μου και για να τα συζητήσουμε αυτά, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να κινηθούμε και ταχύτερα. Για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επάνω στα κείμενα. Και ένα ακόμα θέμα. Μία ερώτηση προς τον κύριο Σέρκας. Τι εννοεί με την συλλογική αυτοαπασχόληση. Προσπάθησα να ε, βρω το νόημα της ορολογίας αυτής, αλλά δεν ήταν σαφής για μένα. Ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένε άλλες τροπολογίες, οι οποίες μου αρέσουν, γιατί κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Μια νέα τέταρτη παράγραφος, για παράδειγμα, στην κατευθυντήρια γραμμή 7, εγώ τη δέχομαι όπως είναι, έτσι εν τέλει, όπως είπα, είναι πολύ καλές, πολύ θετικές οι προοπτικές να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο που να είναι ικανοποιητικό για όλους. Δεν χρειάζεται βέβαια να μπω ε, για την ώρα σε όλα αυτά με λεπτομέρειες, γιατί ούτως ή άλλως θα επαναδιατυπωθούν. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα για συγκεκριμένες διατυπώσεις και προτάσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συνεργάτες <clears throat> ότι μπορούν κάλλιστα να μιλούν με τους ε, βουλευτές τους όταν έχουν κάτι να ρωτήσουν, αλλά δεν θέλω συστηματικά να κάθονται δίπλα τους. Προτιμώ να είναι πίσω, στο πίσω μέρος της όχι δίπλα στους ευρωβουλευτές. Φαίνεται δεν έπιασαν το μήνυμά μου, επαναλαμβάνω οι συνεργάτε, οι βοηθοί των βουλευτών να μην κάθονται δίπλα τους, αλλά στο πίσω μέρος της αίθουσα. Αν χρειάζεται κάτι να ρωτήσουν τον βουλευτή τους, να έρθουν να το ρωτήσουν. Αλλά η θέση του συνεργάτη δεν είναι δίπλα στον Ευρωβουλευτή, είναι πίσω, στο πίσω μέρος αίθουσα. για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών μα. Merci. Madame Harkin, puis Madame euh, Steinruck. Madame... Η κυρία Χάρκιν και μετά η κυρία Thank you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Ολβέιρα δεν είναι εδώ και μου ζήτησε να κάνω κάποιε παρατηρήσει στο όνομά τη και έχω και εγώ κάποιε παρατηρήσει. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Η κυρία Ολβέιρα δυστυχώ δεν ήταν σε θέση να διαβάσει όλε τι τροπολογίε, διότι νομίζω ότι όταν τι έλαβε ήταν ακόμα σε διάφορε γλώσσε, αλλά έχει να κάνει κάποιε παρατηρήσει. Συμφωνεί ότι μέχρι το 2020 η απασχόληση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 75% αντί για το 80% που ε, προτάθηκε στην ΕΚΟΝ. Επίσης ε, δεν συμφωνεί να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων ε, που ζουν κάτω από το επίπεδο τη στόχευση από 25% σε 40% διότι δεν πιστεύει ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Και τέλος, συμφωνεί με την υποχρεωτική δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Όσον αφορά τι δικέ μου παρατηρήσει για την έκθεση, εγώ γενικά στηρίζω τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες που στηρίζουν ε, μεγάλο ποσοστό απασχόλησης, ε, την εκπαίδευση, καλές θέσεις εργασίας κλπ. Ο εισηγητής είπε ότι μπορεί να μην είναι διατεθειμένος ε, να δεχτεί τις επικρίσεις ε, σχετικά με το ε, αίσθημα ιδιοκτησία τη στρατηγική της Λισαβόνα, αλλά εάν δεν το δέχεται αυτό μπορεί ίσως να δεχτεί την τροπολογία 52, όπου μιλώ για, την, για το αίσθημα ιδιοκτησία για τους στόχους του 2020 στα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε στην ακρόση με τον καθηγητή Μόντι χθε. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει να κάνει με την εκμετάλλευση του πλήρου δυναμικού της και ελπίζω να το ε, συμπεριλάβει αυτό και αναφέρεται και στο Flex Security, την ελαστική ασφάλεια. Επίση, συμφωνώ με την ε, τροπολογία 78 και υπάρχουν και κάποιε άλλε τροπολογίε που έχουν να κάνουν με τη βαθμιά απόσυρση ε, των δημοσιονομικών κινήτρων. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του εισηγητή γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά. Επίσης ελπίζω να μπορείτε να στηρίξετε τις τροπολογίες που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, την πρόθεση του επιχειρηματικού πνεύματος ε, και την ε, μείωση της, του διοικητικού φόρτου. Και επίσης υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τη συνέργεια, ανάμεσα, με τη συνέργεια και την μείωση της γραφειοκρατίας. Επίσης, κάποιες τροπολογίες έχουν να κάνουν με την αύξηση συμμετοχής ε, των ηλικιωμένων ε, και των αναπήρων. Ε, επίσης, όσον αφορά την ανεργία των νέων και μια πιο απλοποιημένη προσέγγιση, θα ήθελα να συμπεριλάβω την τροπολογία μου για τα μικροχρηματοδοτικά μέσα και την τροπολογία 98, όπου, όπου αναφέρεστε στους φροντιστές. στους φροντιστές. Αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Στάινρου και κατόπιν η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Ρή που στην αρχή ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές καλές τροπολογίες και πολλές τις οποίες θα μπορέσει να συνδυάσει. Σε κάποια σημεία υπάρχει ανάγκη για συζήτηση για να βρεθούν συμβιβασμοί. Αλλά γενικά βρίσκω θετικό ότι υπάρχει ε, μεγάλη συμμετοχή ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ακουστεί η άποψή μας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Έρη που ε, εμένει στον στόχο της πλήρους απασχόλησης όπως και στο θέμα της ε, καλής εργασίας. Χρειαζόμαστε νέες θέσει απασχόληση, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει dumping στον τομέα των μισθών. Η εκρίζωση τη φτώχεια είναι επίση σημαντική, ε, όπως είναι και η νεολαία. Θα πρέπει σίγουρα να συζητήσουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και θα πρέπει να γίνεται διάκριση. Θα πρέπει να εξετάσουμε ξεχωριστά πώς θα τα πραγματοποιήσουμε αυτά. Σημαντικό είναι επίσης, όπως είπε ο κύριος Έρη και η κυρία Χάρκιν, ότι θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξους συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα πρέπει ε, να ε, επανεξετάζονται. Σημαντικό για μένα είναι να μην σκεφτόμαστε μόνο με στόχο το 2020, αλλά να μην χάσουμε και τον ενδιάμεσο στόχο του 2014. Υπάρχει ανάγκη συζήτηση για να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε σε κοινό δρόμο και αυτό είναι σημαντικό. Ε, τώρα που ξεκίνησε η συζήτηση, ε, εφόσον θέλουμε να μας πάρει στα σοβαρά το Συμβούλιο. Θα πρέπει να επιδιώξουμε μια κοινή γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλισεν και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ δημιουργικοί, πολύ παραγωγικοί, πολύ φιλόδοξοι με τον τεράστιο αριθμό των τροπολογιών μας θα είναι σημαντική πρόκληση για τον κύριο Έρη, για την γραμματεία και νομίζω για όλους μας να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές τροπολογίες. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ. Χρειάζεται να εντοπίσουμε τα στοιχεία που όλοι μας θεωρούμε σημαντικά και στοιχεία στα οποία θέλει να εμείνει ο καθένα από εμά. Οι καλέ θέσει εργασία, οι εξοπλιστέ θέσει απασχόληση αναφέρθηκαν από αρκετού. Θα ήθελα και εγώ να το τονίσω αυτό. Έχουμε μία τροπολογία που ζητά αυτό να είναι ε, <clears throat> μια κατευθυντήρια αρχή σε όλες τις πολιτικές απασχόλησεις. Ε, δεν θα σας ε, εκπλήξει ότι οι πράσινες θέσεις απασχόλησης είναι σημαντικές για μας δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε σε κάθε δεύτερη πρόταση, αλλά βρίσκουμε πολύ σημαντικό να αναφέρονται. Θα πρέπει επίση να το ευθυγραμμίσουμε αυτό με το 2020. Εάν ο κοινό μας στόχο είναι να έχουμε μια έξυπνη συμμετοχική ε, και βιώσιμη οικονομία και αγορά εργασίας, ε, τότε τα θέματα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις κατευθυντήριε μα γραμμές για την απασχόληση. Δεν έχουμε αναφερθεί στην κοινωνική κατευθυντήρια γραμμή υπαριθμών 10. Χαίρομαι που το Συμβούλιο έχει ε, συμπεριλάβει εδώ την φτώχεια. Χαίρομαι που δεν την έχει απορρίψει. Ωστόσο, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά τη συνέχεια για να δούμε ε, πώς θα οριστεί πιο συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να παραμείνει η κοινωνική διάσταση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι σημαντική για τις κατευθυντές αυτές γραμμές. Εχθές είχαμε ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών για τροπολογίες που θα υποβληθούν σε τούτη την Επιτροπή και ελπίζω στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτές τις τροπολογίες. Είναι ισχυρές, φιλόδοξες τροπολογίες και πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας, διότι σε μια γυράσκουσα αγορά εργασίας θα πρέπει όλοι να εργάζονται και θα πρέπει να κάνουμε τις σχετικές προβλέψεις ώστε οι γυναίκες να μπορούν να συνδυάζουν τη φροντίδα των παιδιών με τη δουλειά τους ε, και οι άντρε ε, να μπορούν να συνδυάσουν τη δουλειά τους με τη φροντίδα των παιδιών. Ευχαριστώ κύριο Στομασμάν, κατόπιν ο κύριο Σέρκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Σάμπα Έρη για την ε, έκθεση. Αυτό το λέμε σε κάθε εξηγητή, αλλά εγώ το εννοώ πραγματικά. Έχει ήδη υποβάλει πολλές προτάσεις και έχει καταστήσει σαφές ότι είναι διατεθειμένος να δεχτεί μια σειρά τροπολογιών ώστε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Είναι Ηράκλειο το έργο του, διότι έτσι το η έκθεση έτσι θα γίνει ακόμα πιο μακροσκελής. Ε, πολύ συχνά θέλει κανεί μία έκθεση με ένα πλήρες κείμενο αλλά και μία ε, σύνοψη ώστε να είναι ευανάγνωστη, να συμπεριλαμβάνονται όμως όλες οι διάφορες αποχρώσεις. Είμαι ικανοποιημένος με το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών. Χαίρομαι που έχουν επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, Αναφέρεται στις υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Πιστεύω ότι είναι πολύ βασική βάση. θα πρέπει να είναι δυνατή η εργασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η καινοτομία. Επίσης, ευχαριστώ τον Σαμπαέρη που είπε ότι χρειαζόμαστε μια νέα δομή. Χαίρομαι επίση που οι περισσότερες τροπολογίες έχουν ε, θέμα την αντίσταση στους χαμηλούς μισθούς. Ε, δεν θα πρέπει η ανταγωνιστικότητα να οδηγήσει σε πτώση των μισθών και να μην υπάρχουν ε, ούτε οι ελάχιστες ευκαιρίες στις δομές αυτές και με όλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών, μελών έχουμε διαφορετικά συστήματα ευρέσεως εργασίας, αλλά θα πρέπει αυτά να μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό πραγματικά το βρίσκω σημαντικό. Δεν ε, συμφωνώ πάντα με τους ε, αριστερούς. Ε, να πω όμως για την τροπολογία 120 ότι εδώ αναφέρονται οι κοινωνικοί εταίροι. Εγώ πρόβλημα έχω με την τροπολογία 157 που αναφέρεται στην καλή εργασία. Στην ε, Γερμανία έχουμε πάντα τους καλούς ανθρώπους, τους καλούς ε, πολιτικούς ε, που είναι ενάντια στους άλλους. Εδώ πέρα μιλάμε για τους καλούς εργαζομένους. Χρειαζόμαστε ευέλικτες ευκαιρίες εργασίας που θα πρέπει όμως να έχουν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Η ευελιξία δεν θα σημαίνει ότι μπορούμε να σπρώχνουμε από εδώ και από εκεί τον κόσμο. Η ευελιξία μπορεί να λειτουργήσει όταν υπάρχει ε, αρκετή ασφάλεια. Αυτό το έχουμε συζητήσει και στην Επιτροπή μας ε, με βάση την έκθεση του Όλε Κρίστενσεν. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τη συνάδελφο Στάινμπρουκ ε, για την ε, τροπολογία 148. Πιστεύω ότι η θέση της είναι πολύ σωστή. Αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και λέει πόσο σημαντικό είναι αυτό για τις περαιτέρω ευκαιρίες στην εργασία, να μπορεί κανείς να καταρτίζεται. Θα χρειαζόμαστε λειτουργικές ε, ε, ε, ευέλικτου τρόπου μετάβαση από την μία εργασία στην άλλη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν. καθώς επίσης με τις τροπολογίες 153 και 199 των συναδέλφων Ρία και Σάπα Έρη που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει να απλοποιηθούν πολλά πράγματα. Θα πρέπει όμως να στηρίξουμε, να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διότι αυτό μπορεί πραγματικά να φτάσει τους ανθρώπους ε, που έχουν ανάγκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι σαφής απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει ε, πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ε, είδα κάποιες τροπολογίες των πρασίνων, όπως ε, την τροπολογία 152. Βρίσκω ότι εδώ γίνεται μια εξαιρετική διάρθρωση. Ίσως θα μπορέσει ο Τσαμπαοέρη να την, να την εκλάβει αυτήν ως βάση. Πρόβλημα έχω με την τροπολογία της με αυτό που είπε η συνάδελφο ε, Κορνέλησεν σχετικά με τις πράσινες θέσεις εργασία. Αυτό δεν είναι αίτημα μόνο μιας πολιτικής ομάδας. Έχουμε μάθει πολλά ένας από τον άλλον σε, διάφορες, σε διάφορους σχηματισμούς ε, και οι χριστιανοδημοκράτες ε, είναι υπέρ του να συμπεριληφθούν οι πράσινες θέσει εργασία Δεν θα πρέπει όμω να είναι αυτό σήμα κατατεθέν μια πολιτική ομάδα, Με αυτό διαφωνώ. η συνάδελφο Σρούτερ ε, συχνά φοράει πράσινο φουλάρι και μάλλον έτσι δείχνει τη θέση της. Ε, Μήπω θα πρέπει και εγώ να φοράω πράσινη γραβάτα για να δείξω ότι δεν απέχω πολύ από την ε, άποψη αυτή. Ε, αγαπητέ Σάμπα, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ε, τις επόμενες εβδομάδες ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλού συμβιβασμού, όχι μόνο με του κοινωνικού συζητητές αλλά και με του άλλου, που έχουν υποβάλει πολύ καλές τροπολογίε. καλή διασκέδαση στη δουλειά αλλά νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ, ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Όρι Να απαντήσω και στην ερώτηση που μου έκανε για τις τροπολογίες μου, όπου επανειλημμένως μιλώ για την κοινωνική οικονομία και την αυτοπασχόληση. Κύριε Όρι, συμφωνώ με την προσέγγιση σας και για μια ακόμη φορά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πραγματικότητα. Πάνω από το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στηρίζονται σε μια νοοτροπία και μια αντίληψη περί επιχείρησης που στηρίζεται περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και όχι στο οικονομικό κεφάλαιο. Και σε μια οικονομική κρίση, όλες οι μορφές αυτοαπασχόλησης θα πρέπει να υποστηριχθούν από τις κυβερνήσεις. Μιλήσαμε για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, αλλά επιχειρηματικό πνεύμα έχει κάποιος που αναλαμβάνει τον κίνδυνο, ιδρύει την δική του επιχείρηση για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Αλλά ακόμη πιο έντονο επιχειρηματικό πνεύμα δείχνουν αυτοί που συγκροτούν συνεταιρισμού, σωματεία και δημιουργούν όχι απλώς αυτοπασχόληση, αλλά συνεργάζονται και με άλλους αυτοπασχολούμενους και έτσι καταλήγουμε σε υψηλή προστιθέμενη κοινωνική αξία και κοινοφελείς υπηρεσίες που είναι πολύ κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό κατέθεσα και τις σχετικές τροπολογίες, κύριε Ωρή. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλες οι μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένες και της αυτοπασχόλησης, πρέπει να υποστηριχθούν πολλό δε μάλλον τώρα που διανύουμε μια κρίση γιατί όλες αυτές οι μορφές απασχόλησης έδειξαν ότι είναι πολύ αποτελεσματικές, ώστε να μπορούν τα ίδια τα θύματα της κρίσης να, μπορούν, να μπορέσουν να βρουν κάποια λύση, ξεκινώντας από τους ίδιους. Η, η κοινωνική οικονομία είναι πολύ σημαντική και, και η κοινωνική οικονομία ενισχύεται το να καθένα κάνει τη δική του επιχείρηση, γιατί έτσι είναι που δημιουργούνται εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης και δημιουργείται ένας ενάρετο κύκλος όπου αναβαθμίζεται και το επιχειρηματικό πνεύμα και δίνουμε αξία και στην αυτοαπασχόληση. Γιατί δεν αναφέρεται ότι η κοινωνική οικονομία, ούτε η προσπάθεια να ενισχυθούν τέτοιες πλούσιες μορφές ε, και πολύ ανθρώπινες κοινωνικές μορφές απασχόλησης που και, απο... και οικονομικά είναι και πολύ αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελίν και μετά η κυρία Φιγκερέντα. Ευχαριστώ. Τι κρίμα που Απλώς πρόκειται για διαβούλευση εδώ και δεν μπορούμε να έχουμε την επιρροή στις κατευθυντήρες γραμμές επειδή ξέρουμε ότι έχουν περάσει την ουσία. Παρ' όλα αυτά αξίζει τον κόπο να κάνουμε την προσπάθεια. Θα δείτε και από τις τροπολογίες που έχω καταθέσει, στην 51 μιλώ για τη φτώχεια, στην 60, για τη φτώχεια, συγγνώμη, στην 62 μιλώ για ειδικά μέτρα κατά των διακρίσεων, στην 99 και ούτω καθεξής. Και έχω και την 149 όπου μιλώ ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες για να εξασφαλίσω ότι δεν θα μείνουν ε, απ' έξω από την εξίσωση για να μπορέσουν να προσλάβουν και πιο ηλικιωμένους και έχετε αντιληφθεί ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο προσπαθώ να το περιλαμβάνω παντού. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι πράσινες θέσεις ε, εργασίας ε, είναι σημαντικές, άρα δεν μιλώ μοναχά για μη διακρίσεις οι πράσινες δουλειές πρέπει να μπουν μέσα στο κείμενο και να παραμείνουν. Σωστό. Το άλλο για την μη επαγγελματική κατάρτιση ε, το έχω βάλει στην 241. Αρκούμε σε αυτά, θα συζητήσουμε βέβαια τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκερέντα και μετά ο κύριος Χέντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι ένα έργο που θα γίνει γύρω από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές είναι κολοσιαίο. Γιατί οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άτολμες, αδύναμες, έχουν πολλά κενά και αδυναμίες και μάλιστα επισημάνθηκαν από πολλούς. Για παράδειγμα, θέματα ισότητας ευκαιριών, ισότητας των δύο φύλων, από κοινωνική άποψη υπάρχουν πολλές αδυναμίες, αλλά και μακροοικονομική άποψη υπάρχουν πολλές αδυναμίες, γιατί πολλές φορές κάποιες μακροοικονομικές πολιτικές ήταν η ρίζα του κακού της ανεργίας και της φτώχειας. Γι' αυτό και χρειάζεται ένα τιτάνιο έργο για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Και όπως είπε η κυρία Λίν, Κρίμα που πρόκειται απλώς για μια διαβούλευση και μια σύσταση. Γιατί τον τελικό λόγο στο θέμα αυτό το έχει η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και όχι δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως το έργο είναι δύσκολο και είναι πραγματικά άθλος για τον εισηγητή μας να ολοκληρώσει αυτή την έκθεση. Και αναγνωρίζουμε πραγματικά τις τεράστιες δυσκολίες που εμπεριέχει ένα τέτοιο έργο. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας όχι μόνο στην ανάγκη βελτίωσης της γνωμοδότησης αυτής, αλλά να υπογραμμίσω αυτά που είπε η συνάδελφος Κορνέλισεν. Να ληφθεί υπόψη γνωμοδότηση και της Επιτροπής των Γυναικών που προσπαθεί να συμπεριλάβει και ένα νέο τομέα σε αυτές τι κατευθυντήριε γραμμές και πέραν της οριζόντιας ε, προσέγγισης που έχουμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών που θα πρέπει να περιλαμβάνεται συστηματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτό είναι το mainstreaming, συστηματική συμπερίληψη του θέματος της ισότητας των φύλων σε όλες τις κοινωτικές πολιτικές και επίσης και το κοινωνικό ζήτημα θα πρέπει να αναφέρεται συστηματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να λαμβάνεται υπόψη και του κοινωνικού θέματο θέλουμε ένα mainstreaming. Και επίση ελπίζω να ληφθούν υπόψη κάποιε πιο φιλόδοξες προτάσεις τη δική μου πολιτική ομάδα να δώσουμε ένα μήνυμα για ανάγκη μεταρρύθμιση των πολιτικών. Επίσης, καλό θα ήταν να συζητήσουμε και το άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισαβόνα. Μερικοί το έχουν αποκαλέσει οριζόντια κοινωνική ρήτρα. Αν όμως ήταν πραγματική οριζόντια κοινωνική ρήτρα, η πλειοψηφία των μακροοικονομικών πολιτικών ε, της Ένωσης θα ήταν ε, αντίθετες με τη συνθήκη. Θα ήταν ασυμβίβαστες με τη συνθήκη, γιατί οι περισσότερες μακροοικονομικές πολιτικές της Ένωσης ενισχύουν τη φτώχεια, ενισχύουν ε, την ανεργία, κάτι που αντιβαίνει κατάφορα στο σημείο νέα της συνθήκης. Ευχαριστώ. Κύριος Χέντελ και μετά κυρία Πλάμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία του εισηγητού μέχρι τώρα και τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών δεν τον θεωρώ ως κριτική στην εργασία του εισηγητού, αλλά περισσότερο ως απόδειξη της μεγάλης σημασίας του θέματος. Έχω να κάνω τώρα τα σχόλια. Θεωρώ ότι με την έκθεση αυτή έχουμε μια καλή ευκαιρία να τονίσουμε ότι το ζήτημα της εύκαμπτης απασχόλησης πρέπει να σημαίνει και περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους σε συνθήκες ευκαμψίας. Πρέπει να τονιστεί αυτό. Όσο πιο εύκαμπτη θα είναι η θέση απασχόλησης, τόσο πιο ασφαλής πρέπει να είναι από άποψη εργατικού και κοινωνικού δικαίου. Το ίδιο θα χαιρόμουν αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια κατευθυντήρια γραμμή που να επιγράφεται καλή εργασία. Δεν είναι επινόηση της Ευρωβουλής αυτό. Υπάρχουν αυτά, βελτίωση δηλαδή της κοινωνικής ένταξης και με άλλα ευεργετικά στοιχεία υπέρ του εργαζόμενου, αυτά τα έχουν πει και οι Ευρωπαϊκές Εργατικές Ενώσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να τονιστεί. Το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής. Συχνά, συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει στα κείμενά της για αξιοποιήσιμη εκπαίδευση. Εμείς αξιοποιήσιμη επαγγελματικά δηλαδή. Ε, ε, εμείς όμως δεν θέλουμε μοναχά επαγγελματικά αξιοποιήσιμη εκπαίδευση. Θέλουμε γενικότερα εκπαίδευση που θα είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Αυτά είναι τα τρία αυτά θέματα που θα ήθελα πολύ, αν είναι δυνατόν, να ενταχθούν στις διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε με τον εισηγητή. Η κυρία Πλούμ είναι η τελευταία που έχω σημειώσει εδώ. Ε, μετά θα πω μια φράση εγώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα με την σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Όρη για το πνεύμα συνεργασίας που έχει επιδείξει και είμαι σύμφωνη με την κυρία Λίν. Είναι κρίμα ότι απλώς πρόκειται για διαδικασία διαβούλευσης. Ελπίζω πάντως χάρη στις τροπολογίες καθώς και στις βελτιώσεις που θα επιφέρουμε στο κείμενο της Κομισιόν οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές να αποτελέσουν παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την δημιουργία μιας ομάδας, συγγνώμη, μιας ε, αγοράς εργασίας που να είναι πιο ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Έχω ορισμένες τροπολογίες όπου τονίζω το γεγονός ότι οι χώρες μέλη στον βαθμό που τι σέβονται αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, γιατί έχω ήδη παρουσιάσει την περίπτωση της Ρουμανίας, Έχω τονίσει δηλαδή ότι οι γυναίκες πρέπει να εκπροσωπηθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας. Το ίδιο και οι νέοι. Χαίρομαι που είπατε ότι θα χρειαστεί μια ολοκληρωμένη πολιτική για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ε, εθνοτικών ε, ομάδων, των μειονοτήτων γενικότερα ε, και εννοώ τους Ρωμά κυρίως εν προκειμένου. Χρειαζόμαστε λοιπόν ξεκάθαρες πολιτικές για τον στόχο αυτό. Επίσης πρέπει να καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία και κυρίως μέσα στην οικονομία της κρίσης η οποία κρίση έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρομαι στους τροπολογίες μου και σε πολιτικές που έχουν στόχο να διευκολύνουν τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, προώθησης των, της ενεργού τρίτης ηλικίας, της πρόσβασης των ε, αναπήρων, των μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων, σε τρόπον ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασία όλων, εργασίας όλων αυτών των ομάδων. Επίσης, ας σκεφτούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε τις μονογονικές οικογένειες, που ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως τώρα, αποτελούνται από την μητέρα, συνήθως και πάνω από 90% των περιπτώσεων, αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρότατο κίνδυνο απόλυσης από τις εργασίες τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και εύχομαι να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να συμβάλλουμε σε μια βελτίωση της αγοράς εργασίας τα επόμενα 10 χρόνια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και να επαναλάβω αυτό που είπε και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε το διακύβευμα με τη συγχώνευση των γραμμών, γιατί θέλουμε μια γραμμή για την πολιτική συνοχής. Γι' αυτό ζητήσαμε συγχώνευση. Όταν όμως μιλούμε για πολιτική συνοχής, πρώτα απ' όλα έρχεται στο μυαλό μας όχι τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές. Αν είχαμε μια κατευθυντήρια γραμμή για την συνοχή θα έπρεπε να τη λέμε χωροταξίας περισσότερο γραμμή. Γιατί οι κατευθυντήρες γραμμές δεν είναι μηχανισμός ε, για τη χρήση των κοινοτικών ε, διαδικασιών. Είναι ένας προσανατολισμός περισσότερο. Μία πρόταση για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς. Και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δεν ε, περιορίζονται στην κατανομή των διαφορετικών κονδύλιων. Υπάρχει μια μικρή αντίφαση εδώ πέρα. Καταλαβαίνω την ιδέα του εισηγητού, γιατί μια και οι κατευθυντήρες γραμμές είναι το μέσο εφαρμογής της στρατηγικής του 2020 και στο στρατηγική του 2020 έχουμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης και όταν θα μιλήσουμε για αναθεώρηση των διαρθρωτικών ταμείων, θέλουμε να, να βελτιώσουμε και τη πολιτική συνοχή στα πλαίσια της νέας μεταρρύθμισης, αλλά πώς θα ληφθεί αυτό το στοιχείο στις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση δεν βλέπω. Πώς θα έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή απασχόλησης, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν κάτι στον προπολογισμό. Υπάρχει μια αντίφαση για μένα εσωτερική, δεν μπορώ να καταλάβω. Και όπως είπαμε χθε επ' ευκαιρία της ανακοίνωσης, μετά τη συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους ε, τους επιφορτισμένους ε, με τέτοια θέματα, και το επιτελείο που γνωρίζουμε που θα είναι αυτό που θα διαπραγματευτεί τα τα πράγματα πριν την ε, έγκριση της έκθεσης ε, ορί. Από ό,τι κατάλαβα τους εκπροσώπους των κρατών υπάρχει ένα ανοιχτό πνεύμα ως προς την βασική πρόταση του κυρίου Ορή, δηλαδή το 90% των νέων ε, είτε να προσανατολιστούν προς την αγορά εργασίας είτε προς συνέχιση των σπουδών. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ σημαντική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και θα μπορούσαμε να την έχουμε ως βάση διαπραγματεύσεων για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, γιατί υπάρχει ένα άνοιγμα του Συμβουλίου προς τις τροπολογίες, τουλάχιστον μερικές, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε μια και υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας με το Συμβούλιο και αυτή η διαλλακτικότητα για τα σημεία αυτά, έχετε το υπόψη κατά τη σύνταξη των συμβαστικών σας τροπολογιών. Θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να είμαστε ρεαλιστές για να διαμορφώσουμε μία στεναρή θέση του Κοινοβουλίου και να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο, γιατί άσχετα με τη θέση της εκάστοτε Προεδρίας, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα. Γιατί στις επιστολές μας λένε πολλά και διάφορα ότι η οριστικοποίηση της θέσης του Συμβουλίου θα γίνει μετά την αποκριστάλωση της θέσης του Κοινοβουλίου, αλλά πολλές φορές ε, το Συμβούλιο προχωρεί ερήμην του Κοινοβουλίου. Οπότε καλό θα ήταν εμείς να προτείνουμε δύο-τρεις θέσεις που μας βρίσκουν σύμφωνους και να αποτελέσουν ε, την ισχυρή μας διαπραγματευτική θέση στις συνομιλίες που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για τις παρατηρήσεις τους. Για άλλη μία φορά, ε, είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Να κάνω όμως κάποιες παρατηρήσεις. Ε, αναφέρθηκε το πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ένδια, τη φτώχεια. Μετά την πρόταση της Κομισιόν, το Συμβούλιο θα πρέπει να αρχίσει να αποφασίζει σχετικά με έναν τρόπο μέτρησης της στόχιας. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας, θα πρέπει να το σκεφτούμε προσεκτικά, ώστε όταν τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν για το θέμα αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε τον τρόπο αυτόν στη και είμαστε τη δουλειά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πω στην κυρία Κορνέλησεν ότι φυσικά συμφωνώ με τις ε, πράσινες θέσεις εργασίας και πιστεύω ότι είναι καλή η ιδέα να, να έχουν ε, σημαντική θέση στη στρατηγική του 2020, αλλά όταν μιλάμε για κατευθυντήριε γραμμέ που κατευθύνουν προ κάποια κατεύθυνση ε, σχετικά με τι ε, που θέλουμε να ε, αναλάβουμε, ε, οι κατευθυντήριε αυτέ γραμμέ θα πρέπει να είναι ευανάγνωστε, εύληπτε. Δεν θέλουμε ένα κείμενο δυσανάγνωστο. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορες ιδέες που αναφέρονται στις τροπολογίες και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές, διότι εφόσον συμφωνήσουμε όσον αφορά τις έννοιες, θα είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε ε, και για τη συγκεκριμένη διατύπωση. Όπως είπα, πιστεύω ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός ε, σύγκλησης. Ε, αναφέρθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πράσινες θέσεις απασχόλησης. Ναι, και μπορώ να είμαι και πολύ συγκεκριμένος. Ε, υπάρχει, για παράδειγμα, η τροπολογία 144 που περιέχει πολλά καλά στοιχεία και που ήδη βρίσκεται στον θετικό μου κατάλογο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ε, έναν καλό συμβασμό. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του Αλεχάνδρο, να πω ότι συμφωνώ η αυτοαπασχόληση να αναφέρεται σε κάποιο βαθμό δεν κατάλαβα μόνο τι είναι οι συλλογικές μορφές ε, αυτοαπασχόλησης. Μιλάμε για τις περιπτώσεις όπου αναγκάζεται ο κόσμος να αυτοαπασχοληθεί ή μιλάμε για την ιονή αυτοαπασχόληση. Άνθρωποι δηλαδή που ουσιαστικά είναι μισθωτοί ε, θα πρέπει να φαίνονται ε, σαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αν μιλάμε ε, για την ε, συνάντηση συνεργασία μεταξύ αυτοαπασχολουμένων, ε, αυτό ε, μπορεί να είναι καλό. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με τον όρο συλλογική αυτοαπασχόληση. Α, αν μιλάτε για ε, συνομοσπονδίες, αυτό μπορώ να το δεχτώ. Είναι θετική η ιδέα αυτή. Ε, αν μιλάτε για συνεταιρισμού. Όσον αφορά την ε, ευελιξία και ασφάλεια, το flexicurity. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε εξετάσει επίσης, αλλά... Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Χέντελ και μπορώ να συμφωνήσω, αλλά μήπως η καλή εργασία δεν είναι κατάλληλος όρος, ίσως μπορούμε να βρούμε εναλλακτικό όρο. Δεν έχω πρόβλημα με την ίδια την έννοια, με την ίδια την ιδέα όσον αφορά αυτά που είπε η Πρόεδρος ε, για την ε, συνοχή. Αυτό είναι πιο σημαντικό πρόβλημα και πράγματι αποτελεί σημαντική πρόκληση. Βλέπω να υπάρχει κάποιος κίνδυνος εδώ. Όταν ε, μιλούσαμε ε, για τη δημιουργία της στρατηγικής 2020, ε, μιλούσαμε για τις κατευθυντήρες γραμμές στον δικό μας τομέα. Δεν, μιλούσαμε, δεν συζητήσαμε όμως τις δημοσιονομικές στοιχείες. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς θα χρηματοδοτηθούν οι στόχοι αυτοί. Η πολιτική συνοχής λοιπόν θα πρέπει να οριστεί ή τουλάχιστον ε, να επανακαθοριστεί η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας και προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε. Θέλουμε να έχουμε ε, ε, συμμετοχή και βιώσιμη απασχόληση. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στη συνοχή, θα πρέπει να συζητήσουμε τις οικονομικές κατευθυντήρες γραμμές. Θα μπορούσαμε στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο να πούμε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδέα, αλλά μπορούμε να τη βάλουμε κάπου αλλού στο κείμενο. Μπορούμε να συζητήσουμε διάφορε μορφέ ε, εκπαίδευση. Όπω σα είπα, δεν έχω αντίρρηση ω προ την ιδέα αυτή καθ' αυτή, αλλά θα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τρόπο χρηματοδότηση. Αυτό αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε τους ε, ε, τομείς που δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Θα πρέπει η ε, πολιτική συνοχή να βοηθήσει στην πρόθεση των τομέων αυτών. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον εξοραϊσμό κάποιων πόλεων, το να μορφύνουμε μια πλατεία. Θα πρέπει αυτό να το ενσωματώσουμε στη γενικότερη πολιτική ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε την ιδέα, την έννοια αυτή καθ' αυτή, αλλά απομένει πολλή δουλειά να γίνει. Ούτε λέω ότι θα πρέπει να βιαστούμε να το κάνουμε τώρα αμέσω. Ε, ίσως μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Είμαι διατεθειμένος ε, να συνεχίσω τη δουλειά μου πάνω στο κείμενο τις επόμενες εβδομάδες. Θα προτείνω κάποιες ώρες την επόμενη εβδομάδα στους συναδέλφους... για να δούμε πότε μπορούμε να συναντηθούμε ενδεχομένω σε μικρές ομάδες. Όπως σα είπα ε, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, είμαι ευέλικτο γιατί θέλω να προωθήσω το θέμα. Ε, θέλω κάποια στιγμή να καταφέρω να ολοκληρώσω τη δουλειά, διότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το χρόνο που χρειάζεται για τη μετάφραση των διαφόρων εγγράφων. Οι πολιτικέ ομάδε, θα πρέπει να μπορούν να συζητήσουν τους, ε, τις συμβαστικές προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν ε, σχετικά γρήγορα να καταλήξουμε σε, ε, στη διατύπωση των συμβασμών για να έχουμε τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την υιοθέτησή τους. Ελπίζω λοιπόν την επόμενη εβδομάδα να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε σχετικά με τη συνέχεια του χρονοδιαγράμματος, της πορείας δηλαδή της εκθέσεως, θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε μεταξύ 13 και 14, 14 και 14 Ιουλίου, να διατηρήσουμε την δυνατότητα ενδεχομένω να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα αυτών των δύο ημερών. Αλλιώς έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει η Βελγική Προεδρία για να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε τριμερή διάλογο πριν από τις θερινές διακοπές με την συνεργασία σας να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρονοδιάγραμμά μας. Πάντως, την ψηφοφορία την βλέπω είτε στις 13 είτε στις 14 Ιουλίου μαζί με χρόνο να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Εδώ λοιπόν λύγει το θέμα αυτό. Χθες σας είχα πει ότι ο εκπρόσωπος του ο ΟΣΑ που επρόκειτο να παρουσιάσει μια μελέτη για την εξέλιξη της απασχόλησης στο τοπικό επίπεδο δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσέλθει, άρα θα εξετάσουμε την μελέτη αυτή όταν θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας τον Σεπτέμβριο και σας δίνω ραντεβού για την επόμενη περίοδο των εργασιών μας που όπως σας είπα πριν θα είναι στις 13 έως 14 Εβδόμου.